ερχόμαστε στο, στην διάταξη βάσει του άρθρου 149 της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε το οριστικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης της 20 Ιανουαρίου. Για σήμερα δεν έχω καμία προσθήκη ή αλλαγή για αύριο. Η ομάδα της Ευρώπης των Εθνών και της Ελευθερίας έχει ζητήσει να γίνει μια έκτακτη συζήτηση για την εξάπλωση του ιού Τσιζίκα ως πρώτου σημείου το απόγευμα. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Ζουέλ Μελάν για να παρουσιάσει την αίτηση της ομάδος της Ευρώπης των Εθνών και της Ελευθερίας. Κύριε Πρόεδρε, βάσει του άρθρου 53, καλώς δεχτήκατε αυτή την αλλαγή στην ημερήσια διάταξη. Η ομάδα μας θα ήθελε μια δηλώση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο για αυτήν την επιδημία που τόσο ξαφνικά πλήττει τον κόσμο μας και να ακολουθήσει και συζήτηση στην, στο ημικύκλιο. Λόγω των χαρακτηριστικών αυτής της επιδημίας για την οποία δεν γνωρίζουμε επαρκώς αν είναι απλώς ένας ιικός πυρετός ή εάν ε, μεταδίδεται με τα κουνούπια, θέλουμε να μην έχουμε επανάληψη της καταστροφικής διαχείρισης του θέματος του ιού έμπολα και να μην υπάρξει η ίδια καθυστέρηση που είδαμε να είναι τόσο επιβλαβής ε, εκ των υστέρων. Γι' αυτό, συνάδελφοι, ελπίζω θα συμφωνήσετε. Είναι σημαντικό να συζητήσουμε στο ημικύκλιο το θέμα αυτό και να έχουμε την κατάλληλη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Μελέν. Θέλει κάποιο να υποστηρίξει αυτή την αίτηση, να λάβει το λόγο υπέρ τη αίτηση αυτή. Παρακαλώ. Θέλετε να μιλήσετε θετικά για την αίτηση αυτή. Ήθελα να τοποθετηθώ κατά του αιτήματο, Πρόεδρε. Κύριε Λαβία, πρέπει πρώτα να μιλήσει κάποιος υπέρ. Ο κύριος Ερέρο νομίζω ζήτησε να λάβει το λόγο. Κύριε Γκερέρο, έχετε το λόγο. Ε, κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να παρουσιάσω στην πραγματικότητα μια αναλλακτική πρόταση, λέει ο κύριος Γκερέρο. Όπως είπε η κυρία Μελέν, όλοι δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα για αυτόν τον ιό, ο οποίος διαδίδεται από ένα είδος κουνουπιού και πράγματι αύριο η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας θα μας δώσει πρόσθετες πληροφορίες για την εξάπλωση αυτού του ιού. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα ήταν πιο σόφρον να διοργανώσουμε μια συζήτηση πιο ε, τεκμηριωμένη στην αρμόδια Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που θα μας δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη στιγμή που θα είναι σε επαφή με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Επιμένω, θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο πλήττει πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής. Έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία πολλών ανθρώπων, ιδίως των γυναικών που είναι έγκυες. Υπήρξαν κάποιες περιπτώσεις ήδη ε, εμφάνιση του ιού αυτού στην Ευρώπη και πρέπει η Κομισιόν να αναλύσει το θέμα αυτό ε, και επομένως να επανέλθουμε παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε μια συζήτηση για το ζήτημα αυτό. Εντάξει, λέει ο πρόεδρος. Εν πάση περιπτώσει, εσείς δεν υποστηρίζετε την εγγραφή στην η διάταξη αυτής της έκτακτης συζήτησης. Ποιος είναι υπέρ της πρότασης της κυρίας Μελέν, παρακαλώ. Κατά. Αποχέ. Η πλειοψηφία είναι εναντίον λοιπόν. Και θεωρώ ότι εφόσον έχουμε την έκθεση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας θα πρέπει η αρμόδια επιτροπή να επιληφθεί. Εντάξει. Κύριε Ρέντιν. Για ένα διαδικαστικό, Πρόεδρε με ενημέρωσαν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να εργοποιήσετε το άρθρο 175 για την αναβολή της ψηφοφορίας για το ψήφισμα για τη Συμφωνία ΤΙΖΑ. Θα ήθελα να θέσω υπόψη ότι ο πρόεδρος της ΣΥΝΤΑ, ο εισηγητής, οι σκιώδεις εισηγητές και οι βασικές πολιτικές ομάδες θέλουν να ψηφίσουμε την Τετάρτη θα πρέπει να ψηφίσουμε αυτό το ψήφισμα, διότι είναι καθόλου και τυπικά εντάξει. Αυτό το δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε. Ε, Κυρία Ρέντεν, θα επανέλθω σε αυτό το οποίο ζητάτε. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε καταρχήν το θέμα της παραπομπής στην Αρμόδια Επιτροπή για τον ιό ΖΙΚΑ. Από ό,τι βλέπω η Ολομέλεια υποστήριξε την αίτηση του κυρίου Γκερέρο. Δεν βλέπω να υπάρχει καμία αντίρρηση. Ούτως απεφασίστη να παραπενθεί στην αρμόδια επιτροπή. Κυρία Ρέντινγκ, τώρα εσεί αναφέρεστε σε ένα θέμα το οποίο είναι αργότερα στην ημερησία διάταξη. Αλλά ψηφίστε την Τετάρτη. Εγώ δεν έχω καμία πρόθεση αυτή τη στιγμή να γίνει αναπομπή στην αρμόδια επιτροπή. Από ό,τι γνωρίζω υπάρχουν περίπου 70 τροπολογίες, αλλά ενδεχομένως η, δεν ξέρω πότε εκπνέει η υποθεσμία που είναι απόψε το βράδυ στις 7 ή όχι. Ενδεχομένως θα υπάρχουν και άλλες τροπολογίες ή για διαχωριστή ψηφοφορία. Οι, οι υπηρεσίε του Κοινοβουλίου μου έχουν πει προληπτικά ότι ενδεχομένως θα πρέπει να ληφθεί μια απόφαση σε σχέση με την ε, ε, ψηφοφορία της έκθεσης αυτής. Εγώ πρέπει να σας ομολογήσω ότι δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα ακόμα, ούτε καν προληπτικά. Και δεν έχω καμία πρόθεση, επομένω, όπως λέτε, να αναβάλω την ψηφοφορία. Για πρώτη φορά το αντιμετώπισα το θέμα σήμερα το απόγευμα, μόλις έφτασα όταν μου είπα η υπηρεσία του Κοινοβουλίου ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρξει αναβολή της ψηφοφορίας. Λαμβάνω υπόψη όμως αυτό το οποίο λέτε. Κύριε Βέμπερ Εγώ θέλω να υποστηρίξω αυτό που είπε η κυρία Ρέντινγκ. Αυτή όμως η αίτηση την οποία αναφέρει έχει η πρόταση της κυρίας Ρέντινγκ έχει υποστηριχθεί από την ευρεία πλειοψηφία της αρμόδιας επιτροπής. Μόνο δύο πολιτικές ομάδες θέλουν να επιβραδύνουν και να, κατα... να καταδαπανίσουν χρόνο και να καθυστερήσουν την ψηφοφορία. Επομένως αυτό δεν νομίζω ότι πρέπει να το αποδεχτούμε και δεν αξίζει καν να το συζητήσουμε καταγράφω αυτό που είπατε. σα είπα όμως ότι οι γραμματείε, η γραμματεία μας είπε ήδη ότι υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο γιατί μπορεί να κατατεθούν τέτοιες τροπολογίες οι οποίες έχουν ως στόχο την καθυστέρηση. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν όμως και τροπολογίες οι οποίες είναι ε, τυπικά έγκυρες και είναι τροπολογίες ουσίας. Εάν είναι πραγματικά τροπολογίες μόνο τυπικού χαρακτήρα δεν είμαι υποχρεωμένος να τις αποδεχτώ. Ως πρόεδρος και η αρμόδια αντιπρόεδροι όταν γίνεται μία ψηφοφορία δεν, ε, δεν κάνουμε αυτόματα την αναπομπή ε, των εκθέσεων ακόμα και όταν έχουν 300 ή και παραπάνω τροπολογίες. Πολλές φορές λοιπόν Υπάρχουν πολλές ε, διαμαρτυρίες των βουλευτών για το ότι δεν κάνουμε αναπομπή στην αρμόδια επιτροπή. Ξέρω ότι έχει ε, επιληφθεί του θέματος αυτού η Επιτροπή Συνταγματικών Θεμάτων, γιατί αυτό είναι πραγματικά σημαντικό θέμα για τον κανονισμό του Κοινοβουλίου. Κόρμπετ. Πράγματι, Πρόεδρε, όμως το άρθρο 175 δεν ε, αφορά την αναπομπή ενός θέματος στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Απλώς ζητά όταν υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός τροπολογιών, η Επιτροπή αυτή να ε, δράσει ως φίλτρο, ιδίως όταν έχουν υποβληθεί πολλές τροπολογίες που δεν πρόκειται να υιοθετηθούν από την Ολομέλεια. Έχουμε εξετάσει λοιπόν το θέμα και είδαμε ότι το 1 δέκατο τουλάχιστον των τροπολογιών δεν πρόκειται να περάσουν. Αυτό όμως θα συντομεύσει πάρα πολύ και τη διαδικασία της ψηφοφορίας στο σώμα μας. Διότι ήδη θα έχουν περάσει από την ε, κρίση της Επιτροπής οι τροπολογίες. Οπότε αυτό θα έπρεπε να διευκολύνει τη διαδικασία εάν θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτό το άρθρο. Κύριε Κόρμπετ, θα ήταν ε, χαρά μου να συμφωνήσω μαζί σας. Όμως, έχουμε δει στις δικασίες των Επιτροπών 10% των μελών μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής να αρκούν για να στείλουν τελικά το πακέτο λίγο πολύ απαράλλαχτο ως την Ολομέλεια. Αυτή είναι η εμπειρία μου από τα προηγούμενα χρόνια. Και νομίζω ότι αυτό ισχύει και για την Επιτροπή ΑΦΚΟ, όπως και για τις υπόλοιπες Διαδικαστική παρέμβαση πάλι. Κύριε Φέρα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συζήτηση για την συμφωνία ΤΙΖΑ είναι το ίδιο σημαντική όπω και αυτή για τη συμφωνία TTIP. Δεν μπορείτε να υπερβαίνετε το ρόλο σα. Θέλετε να μα επιβάλλετε μια παροδία τροπολογιών, κάτι που θα θέσει σε κίνδυνο την δημοκρατία του ίδιου του Κοινοβουλίου. Υπάρχει η κοινοβουλευτική ελευθερία εδώ. Και γι' αυτό σα παρακαλώ να σέβεστε το ίδιο και τα κείμενα και του βουλευτέ. Μάλιστα, ευχαριστώ. Ερχόμαστε στο επόμενο σημείο την Τρίτη υπάρχει μια αίτηση της συνομόσπονδης ομάδας των ε, αριστερών που ζήτησε η δήλωση του Συμβουλίου και της Κομισιόν για την αυξανόμενη ε, ξενοφοβία και βία εναντίον ε, προσφύγων να προσθεθεί ως τέταρτο σημείο στην κοινή συζήτηση για την κρίση των προσφύγων, για τον σεβασμό, για τη μη απόθεση και την ε, διευκόνιση για την Τουρκία. Η κυρία Τσίμερ θα αιτιολογήσει αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Έχετε ήδη αναφέρει το περιεχόμενο της αίτησή μας. Μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει το κύριο αυτό σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ιδίως στη Στοκχόλμη, έχουν δημιουργήσει, έχουν δημιουργήσει μια διεθνή ε, προσοχή για τα θέματα των προσφύγων. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πολλές φορές έχουν πολλά παιδιά και βρίσκονται ουσιαστικά υπό δίωξη. Υπήρξαν επιθέσεις εναντίον ε, καταβλισμών και οικειών όπου βρίσκονται πρόσφυγες στην Γερμανία. Ξέρετε ότι επίσης στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις αυτό το τελευταίο Σαββατοκύριακο υπήρξαν ε, διαδηλώσεις ε, ακροδεξιών κατά των μεταναστών και επιθέσεις και κατά τη δική μας άποψη αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να προσθεθεί στην κοινή συζήτηση που θα γίνει την Τρίτη το απόγευμα παρουσία του Συμβουλίου και της Κομισιόν. Και η ομάδα μου, όπως έχουμε αναφέρει, έχουμε ζητήσει μια ονομαστική κλίση για την αλλαγή αυτή της ημερησίας διάταξης. Ακούσατε την άποψή της κυρίας Τσίμερ, ποιος υποστηρίζει αυτή την πρόταση. Κύριε Γκερέρο. Θέλω να υποστηρίξω την αίτηση της κυρίας Τσίμερ, συμμερίζομαι τις ανησυχίες της και θέλω να προσθέσω ότι παρά το γεγονός ότι δεν αναφέρεται ως ειδικό σημείο στην αυριανή συζήτηση του απογεύματος ή δυνατόν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα των χιλιάδων παιδιών που έχουν εισέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή τη στιγμή είναι άγνωστη η τοποθεσία στην οποία βρίσκονται. Είναι αγνοούμενα δηλαδή αυτές οι χιλιάδες παιδιών. Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στην κοινή συζήτηση που θα κάνουμε αύριο το απόγευμα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κάποιος θέλει να λάβει το λόγο κατά της πρότασης της κυρίας Τσίμα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ και πολλά χρόνια ζητάμε να γίνει συζήτηση για τη βία από την ε, που συνδέεται με τα θέματα των προσφύγων. Θέλουμε να συζητήσουμε για όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη βία που περιστρέφεται γύρω από το θέμα των προσφύγων. Είναι άδικο για τις χιλιάδες των θυμάτων, για τις γυναίκες στην κολονία να υπάρξει μια τέτοιου είδου συζήτηση, γιατί υπάρχουν άλλα θέματα τα οποία ζητήσαμε να συζητηθούν και έχει απορριφθεί κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ε, Ερχόμαστε στην ψηφοφορία, λέει ο πρόεδρος. Έχει ζητήσει η κυρία Τσίμερα ονομαστική ε, κλίση και έγινε γέρος και προθέσμος αυτή η αίτηση. Ξεκινά, ξεκινά λοιπόν η ψηφοφορία, η ονομαστική κλίση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. ...183 υπέρ, 142 κατά. Η αίτηση λοιπόν αυτή γίνεται δεκτή. Κυρία Μπέρας, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήθελα να σας πω ότι ε, να επισημάνω ότι ήθελα να υπερψηφίσω αλλά έχω ξεχάσει την κάρτα μου. Μάλιστα το σημειώνουμε στα πρακτικά. Ευχαριστούμε. Έτσι έχουμε οριστικοποιήσει την ημερησία διάταξη για αυτή τη βδομάδα. Ερχόμαστε λοιπόν στο πρώτο σημείο της ημερησίας διάταξης. Είναι η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ο κύριος Μαριάς είναι ο συντάκτης, είναι ο εισηγητής και θα ήθελα με την ευκαιρία